Να φέρουμε μόνο στο Ευρωκοινοβούλιο σε αυτή την περίπτωση. Προχωράμε. Περνάω στα πρακτικά της 25ης Φεβρουαρίου. Έχουν διανεμηθεί. Έχετε τυχόν ερωτήσεις σε σχέση με τα πρακτικά. Εάν όχι, εγκρίνονται. Έχω και μια δήλωση που θα ήθελα να κάνω. Με ενημέρωσαν οι αρμόδιες πολωνικές αρχές